Δεύτερη ανακοίνωση σε σχέση με τις δύο συστάσεις αποφάσεων από πλευράς ε, της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και Μεταφορών ε, προτάθηκε να μην προβληθεί η αντίρρηση, η αντίθεση στη κατεξοδότηση πράξη που ε, ανακοινώθηκαν εχθές στην έναρξη της συνεδρίασης. Δεν κατατέθηκε καμία αντίρρηση μέσα στο 24ωρο που είναι η προθεσμία και σύμφωνα με το άρθρο 87α εδάφιο 6 θεωρούνται εγκριθήσεις οι δύο αυτές συστάσεις, οι οποίες και θα δημοσιευθούν ως ε, τμήμα των κειμένων που εγκρίθησαν αύριο μέρα Τετάρτη. Ακολουθεί τώρα η έκθεση της κυρίας Δελβό και του κυρίου Σιμάνσκι σχετικά με το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό οριζόντα.